Έχουμε και κάποια άλλη ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές της Σουηδίας επικοινώνησαν με τον ε, πρόεδρο και ανακοίνωσαν την εκλογή του κυρίου Γιάκοπ Νταλούντε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κύριο Πίτερ Έριξον, κάτι το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τις 7 έκτου του 16. Καλώς όρισε ο νέος συνάδελφος και σας υπενθυμίζω ότι θα είναι πλήρως ε, μέλος του Κοινοβουλίου και θα συμμετάσχει σύμφωνα με τον κανονισμό σε όλα τα όργανα του Κοινοβουλίου μας.